τι συνέβη. Ευχαριστούμε κύριε Βούρτς για αυτή την πληροφορία. Οπότε θα σκεφτούμε ακόμη πιο σοβαρά και την σφοφορία που θα γίνει αμέσως. Λοιπόν, Ξεκινάμε με την κοινή θέση Συμβουλίου της Αιτιολογήσης ε, και την κοινή θέση του Συμβουλίου. Ο τίτλος θα δημοσιευτεί στα σημερινά πρακτικά. Οπότε από αύριο ξεκινάει η τρίμηνη προθεσμία του Κοινοβουλίου από τις 16 Ιανουαρίου 2009. Ανακοινώνω επίσης πως τα μέλη Μαρτοκαπάτο Κουμπίτσκα, Τόμας μακτάνο και Χέλγκα Τρούπελ κατέθεσαν την ε, γραπτή δήλωση 26 του 2008 για την ε, εκπομπή του σταθμού TDTV στην ε, Κίνα κάτι το οποίο θα διαβιβαστεί σε αυτούς που οποίους σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού και θα δημοσιευτεί στην συνεδρίαση του Φεβρουαρίου 2009. Τον λόγο σχετικά και ο κύριος Καπάτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματος όσων ε, ξεκίνησε την ε, συμβιβαστική αυτή λύση τους υπόλοιπους 440 βουλευτές που συνυπέγραψαν το κείμενο. Εμεί ζητάμε από την UTSAT να ξαναρχίσει τις εκπομπές της MTTV στην Κίνα